Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, good afternoon. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να σας καλωσορίσω στη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Γιατί να καλωσορίσω την Επίτροπό μας την κυρία Γιούροβα για μια ακόμη φορά, θα, μάλλον αργότερα θα σας ξανακαλωσορίσω αλλά αρχικά να εγκρίνουμε παρακαλώ την μερίσια διάταξη με τις εξής αλλαγές στο αρχικό σχέδιο. Το σημείο 5, ψηφοφορία επί του συμπεφωνηθέντος κειμένου για την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών, κυρία Γκέριγκερ ήταν η συγγήτρια, θα μετατεθεί για αύριο, μετά την συνεδρία σκεκρισμένων των θυρών. Η ψηφοφορία τη της Ροζιέρ για την ε, προστασία γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα το σημείο 7 αναβάλλεται όπως και η ψηφοφορία της εκθέσης του κ. Καρύμ για την επικουρικότητα και αναλογικότητα σημείο 8. Επιθυμεί κάποιο ε, να υποβάλει κάποιο αίτημα για αλλαγή στην διάταξη ή θέλει να προβάλλει κάποια αντίρρηση. Όχι. Άρα εγκρίνεται η μερσιά διάταξη με αυτές τις αλλαγές. Θέλω πρώτα να σας παρακαλέσω να βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας γιατί στις 4 αλλά και αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε. Έγκριση των πρακτικών, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης και 16ης Ιουνίου του 2015 θα εγκριθούν. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο σημείο 4 Έχω την τιμή να υποδέχομαι την Επίτροπο κυρία Γιούροβα στο πλαίσιο του διαθρωμένου διαλόγου. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων, συνεργασία του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω στον τομέα της δικαιοσύνης διαφοροποιήθηκε κάπως τα τελευταία χρόνια. Λόγω μια διαφορετική προσέγγιση ό,τι αυτή την νομοθεσία μας ε, υποσχέθηκαν από την Κομισιόν ότι θα έχουμε πολύ λιγότερε νομοθετικέ προτάσει σε σχέση με αυτέ που είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον. Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Υπήρξαν θετικέ εξελίξει όπω τη συμφωνία για τον κανονισμό περί αφαιρεγκαιότητας και βέβαια είχαμε και επιτυχίες τριμερείς διαλόγους ε, για την μεταρρύθμιση της διαδικασίας ε, μικροαξιώσεων που θα την εγκρίνουμε αύριο, τις μικροδιαφορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση για την πρόταση στα δημόσια έγγραφα θα ολοκληρώσουμε την επόμενη εβδομάδα και σε ό,τι αφορά νέες προτάσεις βέβαια περιμένουμε με ανυπομονησία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού Βρυξελών 2 Γνωρίζετε επίσης ότι η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ε, θέσπιση κατώτατων ε, προτύπων για τις αστικές διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο δίνοντάς της τον λόγο. Καταρχάς θα μας παρουσιάσει τις δικές της απόψεις και εν συνεχεία θα ακολουθήσει μια πλήρη συζήτηση. Κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε ε, τη ευρωπαϊκή επιτροπή για το επόμενο έτο. Πριν δούμε το μέλλον όμω, ας ε, δούμε το πρόσφατο παρελθόν πρώτα. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γιούρη και ιδίω ε, την εισηγήτρια κυρία Γκέρνγκερ, Ντέντεμπερκ, όπω και του κοιόδης εισηγητέ και τον κύριο Μπούντα όλο ιδιαίτερο για το συμβιβασμό για αυτή τη διαδικασία σχετικά με τι μικροδιαφορέ. Η ψηφοφορία θα γίνει μετά την ανταλλαγή απόψεων και αποτελεσματικό και αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός θα βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για διασύνοριακές, αστικές και εμπορικές υποθέσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Με βάση αυτή την επιτυχία τώρα πρέπει να προχωρήσουμε να λύσουμε και όσα ζητήματα εκκρεμούν. Είμαι αισιόδοξη ότι σύντομα θα δούμε πρόοδο και σε ό,τι αφορά την οδηγία για την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Βλέπω θετική να είναι δυναμική στο Συμβούλιο και με τη δική σα υποστήριξη θα συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά για να πείσω αυτού που δεν έχουν ακόμη πιστεί, τα αναποφάσιστα δηλαδή ακόμη κράτη-μέλη, να στηρίξουν αυτή την οδηγία. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου είναι αποφασισμένη, ε, είναι δυνατή μια γενική προσέγγιση για το Συμβούλιο του Οκτωβρίου και σε συνέχεια αυτού μπορούμε να ξεκινήσουμε τριμερείς διαλόγους και να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτό θα είναι μια καλή είδηση για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρότασή μας περί απλούστευσης ε, της ε, αποδείξης δημόσιων εγγράφων, οι πρώτες τεχνικές συζητήσεις ε, πραγματοποιήθηκαν ήδη και έχει προγραμματιστεί και ο πρώτος τριμερής διάλογος. Θα λάβει χώρα σε δύο ημέρες. Πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι και να φροντίσουμε να περικοπεί η, απαραί... η μη απαραίτητη γραφειοκρατία, γιατί αυτό θα διευκολύνει τη ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών. Ο προτινόμενος κανονισμός ε, θα ε, καταργήσει την επισημείωση της ε, Χάγης, αλλά πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να έχει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογή. Ε, καλό είναι τα βασικά έγγραφα να παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογή της επιχείρησης, ιδίω τα έγγραφα τα οποία να φέρουν την νομική μορφή της επιχείρησης και ποιο είναι ο εξωτημένος αντιπρόσωπος της επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα χαρά με το Κοινοβούλιο και τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία για να έχουμε ευτυχή κατάληξη μέχρι τα τέλη του έτους και σε αυτή νομοθετική πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προτινόμενο κανονισμό ε, για τις, ε, τα διάφορα καθεστώτα ε, γάμου και άλλων μορφών συμβίωσης, το Σεπτέμβριο έχουμε αποφασίσει να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτά τα συμβαστικά κείμενα και να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο μέχρι το 2015 για να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να επιτύχουμε ομοφωνία, όπω απαιτείται. Εργαζόμαστε σκληρά μαζί με την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου για να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την δέσμευση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ενέκρινε την έκθεσή σα για πρόταση αναθεώρηση ε, τη οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Είναι μια πρόταση σημαντική, ε, μια σημαντική συμβολή για να βελτιώσει την τόσο απαραίτητη διαφάνεια στον τομέα αυτό. Η συζήτηση στην Επιτροπή σας έμαθα ότι ήταν δύσκολη και είμαι πολύ ευγνώμων προς τον κύριο Κοφεράτη, τον εισηγητή, αλλά και όλους τους και τις εισηγητές για το σκληρό έργο που επιτέλεσαν για να επιτύχουν αυτό το συμβιβασμό. Είναι μια πολύ καλή βάση διαπραγματεύσεων. Ομοίως, Ελπίζω να καταλήξατε σε μια καλή συμβιβαστική πρόταση για την πρόταση περί μονοπρόσωπης εταιρείας ΕΠΕ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση και για εμένα, γιατί ουσιαστικά θα απελευθερώσει το δυναμικό της ενιαίας αγοράς για τις μετριόμενες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει οι διαφορές στα εθνικά εταιρικά δίκαια να περιοριστούν όπου μπορούμε βέβαια. Και θα πρέπει να θαρρύνουμε τους επιχειρηματίες να επιλέγουν ε, την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στην πρώτη σε αυτή αναλύονται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, καταχώρηση, τη λειτουργία των ε, εταιριών αυτών ε, στα κράτη-μέλη. Θα έχουμε επίσης ένα υπόδειγμα online. Θα μπορεί να ξεκινήσει μια εταιρεία με κεφάλαιο ενός ευρώ και με απόλυτη ασφάλεια βασικές αρχές και σας ζητώ να τις εξετάσετε. Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δραμική καταχώρηση των ανατεριών, θα βοηθήσει. Έχουμε και την ψηφιοποίηση, ε, έναν ε, κανονισμό που συνάδει με τον κοινό μας στόχο να απελευθερώσουμε το δυναμικό της ενέας ψηφιακής αγοράς πιστεύω ότι ο συμβιβασμός του Συμβουλίου προσφέρει πηδοφόρες λύσεις σε πολλά από τα θέματα που έχει θέσει το Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, 16 κράτη-μέλη ήδη έχουν αυτή την ε, online καταχώρηση και έχουν αξιοποιήσει την εμπειρία του στις συζητήσεις του Συμβουλίου για τη δημιουργία των ασφαλιστικών δικλείδων. Το Συμβούλιο επίσης ήδη προέβησε σημαντικές διευκρινήσεις, Μετοχή των εργαζομένων, resulting from the anti-money laundering directive have to... Και εργασιακοί νόμοι θα παραμείνουν ως έχουν, δεν θα επηρεαστούν. Το θέμα της έδρας ε, ήταν επίμαχο και έχει βγει από το κείμενο. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν επ' αυτού. Θα μπορούν δηλαδή, όπως και τώρα, ελεύθερα τα κράτη-μέλη είτε να επιτρέπουν είτε να μην επιτρέπουν ε, το διαχωρισμό των εδρών. Φαντάζομαι ότι όπω και για μένα και για εσάς είναι σαφέ ότι μεσοπρόθεσμα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό των εδρών. Επίση θα ήθελα να αναφέρω πολύ σύντομα το μηχανισμό, ε, την οδηγία μάλλον για εναλλακτικό μηχανισμό επίλυση διαφορών. 9 Ιουλίου περιμέναμε φέτο να έχουμε ολοκληρώσει από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχουν φτάσει όλα αυτά σε αυτό το σημείο. και θέλω να, ε, το έχω πράξει να επενθυμίσω ε, στους Υπουργούς Δικαιοσύνης ε, τη σημασία αυτού του προγράμματος, αυτού του σχεδίου για, την, για το ODR, την online επίλυση διαφορών. 9 Ιανουαρίου 2016 θα πρέπει να είναι επιχειρησιακός αυτός ο μηχανισμός και ελπίζω τα σημεία επαφή του ODR να καλύψουν τουλάχιστον 50% του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τότε. Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφή ε, δημιουργείται και για να βοηθήσει του εμπόρου, του πολίτε την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αυτοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή. Καταλαβαίνω ότι στι περισσότερε χώρε μέλη η εμπειρία των κέντρων καταναλωτών ε, θα αξιοποιηθεί σε αυτά τα εθνικά σημεία επαφή γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος είναι η αφαιρεγκαιότητα, η σχετική δηλαδή οδηγία. Ο σχετικός κανονισμός, αναδιατύπωση λοιπόν του κανονισμού για την αφαιρεγκαιότητα που αφορούσε το εφαρμοστό δίκαιο, αναγνώριση, εφαρμογή των αποφάσεων, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα παρόλα αυτά. Είχαμε την εκθέση των πέντε Προέδρων πρόσφατα που δείχνει ότι επί της ουσίας εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές στο δίκαιο φερικιώτης των κρατών μελών. Και είναι μια συμφόρηση που δεν επιτρέπει την ενοποίηση των κεφαλαγόρων. Γι' αυτό εξετάζει η Κομισιόν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων και προβαίνει και σε μια συγκριτική μελέτη των ε, εθνικών διαδικασιών αφαιρεγκαιότητα που δεν καλύπτονται, οι πτυχέ δηλαδή που δεν καλύπτονται από τη σύσταση περί αφαιρεγκαιότητα. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και μελέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει ποιο είναι το καταλληλότερο νομικό μέσο για να αντιμετωπίσει τι διαφορέ. Δεν ξέρω πόσο πολύ προσφυλές είναι σε εσά το θέμα της προστασίας οικογενειών και παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή ε, του κανονισμού Βρυξελών 2 και θα καταλήξω σε μια αναθεωρημένη πρόταση την οποία θα σας παρουσιάσω στο πρώτο εξάμεινο του 2016. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν λήψεις ε, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τους υπουργού την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του Συμβουλίου οι διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές ε, πολλές φορές καθυστερούν, πολύ χρονοβόρες διαδικασίες σε ορισμένα κράτη-μέλη, γι' αυτό και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες και να άρουμε ε, τα εφιστάμενα εμπόδια για την αναγνώριση και βολή εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την επιμέλεια των παιδιών. Η, η αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξελών 2α θα πρέπει να βασίζεται και να βελτιώνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν έχουν όλα τα νομικά συστήματα επαρκή διαδικασία εκτέλεση αποφάσεων, λαμβάνοντα υπόψη που να λαμβάνουν υπόψη τι ιδιαίτερότητε των γονικών θεμάτων και διαφορών. Υπάρχουν διαφορέ και στους εθνικούς νόμους ό,τι αφορά την ακρόαση των παιδιών, για παράδειγμα. Ε, πολλές ε, χρησιμοποιούνται για να αρνηθούν να γίνει άρνηση τη εκτέλεση. Ε, ε, απόφαση ξένων δικαστηρίων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση προς συμφέρον των παιδιών. Τέλος. Ε, τον επόμενο χρόνο θα ασχοληθούμε πολύ με τη στρατηγική ενιαία ψηφιακή αγορά. Στόχο της Κομισιόν είναι το να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό στις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή αγορά ε, από πλευρά των Ευρωπαίων καταναλωτών για να απελευθερωθεί πλήρως το δυναμικό της έννοιας ε, ψηφιακής εσωτερική αγοράς. Πολύ λίγοι ε, καταναλωτές αυτή τη στιγμή ψηφίζουν, ε, αγοράζουν ε, μέσω του ίντερνετ ε, ηλεκτρονικά και λίγες επιχειρήσεις σχετικά προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του ίντερνετ. Πρέπει εμείς από τη μεριά μας ε, να ασχοληθούμε με το ενοχικό δίκαιο. Ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να βαρύνονται με πρόσθετα κόστη συναλλαγών ούτε να αντιμετωπίζουν νομική αβεβαιότητα εξαιτία της διαφοράς μεταξύ του ενοχικού δικαίου στις διάφορες χώρες μέλη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δείξουμε στους καταναλωτές την προστιθέμενη αξία της ενιαίας αγοράς ε, που θα πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ε, ετοιμάζουμε νομοθετική πρόταση για εναρμόνιση των κανόνων των επιγραμμικών αγορών ε, βασικά ε, βασικές ρήτρες, ε, συμβατικές ρήτρες για συναλλαγές μέσω διαδικτύου και θεωρούμε ότι τέτοιες προτάσεις είναι πιθανό να ε, ε, εγκριθούν, αλλά μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί το, σύστημα, ε, το επιγραμμικό σύστημα με το ε, σύνηθες μη ηλεκτρονικό σύστημα. αυτό όμως θα προκύψει σταδιακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διασφαλίσει ήδη ε, ενιαίους ε, κανόνες συμβάσεων ε, για θέματα όπως οι πληροφορίες πρώτης υπογραφής ή το δικαίωμα της, ε, ε της απόσυρση, ε, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και άλλα θέματα, όπω θέμα των αποζημιώσεων σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων που ε, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Θέλουμε να εναρμονίσουμε ιδιαίτερα τους κανόνες ε, που αφορούν τα υλικά αγαθά καταναλωτού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λατωματικά ψηφιακά προϊόντα. Θέλουμε να είμαστε όσο το πιο ανοιχτοί και διαφανείς γίνεται στη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της ε, πρότασης και θα μιλήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, γιατί πρέπει να νομοθετήσουμε σωστά στην έκθεσή σας για τον, για τον κοινό ευρωπαϊκό νομοπολίσεων ε, σωστά υπογραμμίσατε ότι το επιγραμμικό εμπόριο είναι η βασικότερη πρόκληση για το μέλλον. Θα χρησιμοποιήσω την εμπειρία σας και θα συνεργαστώ μαζί σας σε αυτή την καινούργια μας πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν οι ερωταπαντήσεις ε, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω την κυρία Μαγκίνες που είναι ο διαμεσολαβητής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγωγή παιδιών. που νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα ε, να θέσουμε και ερωτήσεις τώρα. Η κυρία Ρίγνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Επίτροπο για όλα αυτά που μας είπατε. Ήδη την περασμένη χρονιά μπορέσαμε να συνεργαστούμε και πλέον είναι απόλυτα σαφές ε, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Και έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα, μιλήσατε για το δίκαιο, το πτωχευτικό δίκαιο και επίσης ε, μιλήσατε και για την προσπάθεια να πλησιάσουν λιγάκι και να αρμονιστούν οι σχετικές διαδικασίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να δείτε λιγάκι τις διατάξεις, εθνικές διατάξεις αυτών των, ε, αυτού του πτωχευτικού δικαίου γιατί σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχει ουσιαστικά επεξεργασμένο δίκαιο. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή κατά την άποψή μου η Κομισιόν να επιληφθεί αυτού του θέματος. Και έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα στην Ισπανία κυρίως, όπου έχουμε ένας, έναν ιδιοκτήτη, μία ιδιοκτήτρια σπιτιού, που έγινε μάλιστα και δήμαρχος, δήμαρχος Βακερλώνης ε, και εκρεμεί εις βάρος της μία περίπτωση ε, πτωχευτικού, πτωχευτικού δικαίου, πτωχευτικής περίπτωσης. Το άλλο που θέλω να φέρω είναι Women on Board, οι γυναίκες στα εποπτικά συμβούλια. Ε, να δείτε λιγάκι τις διατάξεις που αφορούν στις γυναίκες που εργάζονται σε υψηλές θέσεις, σε εποπτικά συμβούλια. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως βουλευτές έτσι ώστε να πιέσουμε το θέμα από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Λουξεμβούργου γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και όχι μόνο τεχνικής φύσης θέματα. Τώρα για τα δικαιώματα των μετόχων. Έχουμε εισηγητή, τον κύριο Κοφεράτη, που πιστεύω ότι θα αναφερθεί επί του θέματος. Βλέπετε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό, παρακαλώ να το μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ότι δηλαδή υπάρχει ένα συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέταρτο και πιο σημαντικό θέμα για μένα είναι οι μονοπρόσωπες εταιρείες, single member company. Μιλάτε μόνο για την ψηφιακή καταχώρηση εταιριών. Το single member company, αυτές οι μονοπρόσωπες εταιρείες δεν το χρησιμοποιείτε εύκολα, είσαστε πολύ επιφυλακτικοί επ' αυτού. Παρακαλώ όμως να προσέξετε πολύ το τι ακριβώς μπορεί να γίνει, γιατί στην περίπτωση αυτή όταν πρόκειται για την ψηφιακή καταχώρηση υπάρχει και ο διάβολος στις λεπτομέρειες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λεπτομερείς και ακριβείς κανόνες. Και θέλω να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε όσον αφορά την διασύνδεση των επιχειρηματικών, των εταιρικών μητρώων. Νομίζω ότι εκεί υπολείπονται αρκετά. Και εδώ θέλω επίσης να σας πω κατά πόσον έχετε δει τη 14η οδηγία. Είναι η αιτία του κακού. Είναι η οδηγία που αφορά στη μετεγκατάσταση των εδρών κυρίως. Έχουμε λοιπόν ε, προβλήματα που έχουν προκύψει με τις ε, μονοπρόσωπες εταιρείε και έχει διαπιστωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν ικανοποιητικές διατάξεις για τη μεταγκατάσταση της έδρας μιας επιχείρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι μπορεί να προτείνει αρκετά έτσι ώστε να ξεφύγουμε λιγάκι από τις μονοπρόσωπες εταιρείε. Να ε, σας κάνω μερικές ακόμα ερωτήσεις κύριε Επίτροπε. Κύριε Σάνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, Ευχαριστώ πολύ για την πολύ λεπτομερή αυτή περιγραφή των δραστηριοτήτων σας και των προτεραιοτήτων σας. Ε, δύο θέματα θέλω να θίξω, τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πρώτον, η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου από τον περασμένο μήνα για την αναγνώριση ορισμένων επίσημων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν άτομα που μετακινούνται συχνά από το ένα κράτος μέλος σε άλλο και αυτή τη στιγμή χάνουν πολύ χρόνο προκειμένου ε, να σφραγίσουν και να βεβαιώσουν το γνήσιο των ε, διαφόρων εγγράφων. Το Συμβούλιο υποσχέθηκε πρόοδο. Όμως, περιόρισε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εξαιρώντας πολλά από τα έγγραφα που είχε προτείνει η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν μόνο τέσσερις πολύγλωσσες ε, φόρμες ε, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται με πληρωμή, με κόστος. Ποιο είναι η άποψη της Κομισιόν για την απλοποίηση σε αυτόν τον τομέα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το φόρμ για τα δικαιώματα των παιδιών, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις ε, κακές πρακτικές ορισμένων δικαστηρίων που επιτρέπουν υιοθέτηση χωρίς συγκατάθεση των βιολογικών γονέων. Αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα μεικτά ζευγάρια που προέρχονται δηλαδή από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι ε, φαίνεται η οι, ε, οι ε, ξένοι γονείς που προέρχονται από εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λιγότερα δικαιώματα, έχουν χαμηλότερο στάτου από αυτού που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσει την εφαρμογή της ε, Σύμβασης Βρυξέλλες 2. Ελπίζω ότι η μελλοντική τροποποίηση της ε, συνθήκη αυτή θα το λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Mrs. Hautala. Κυρία Χάουταλα, Επιτροπέ, δύο Τσούλες. Ε, είμαι μόνιμη εισηγήτρια για το Γενικό Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο. Και όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό, όπως επίση και ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ε, ζητούν ε, να υπάρχει ένα τέτοιο, ένα τέτοιο ενοποιημένο διοικητικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο λοιπόν, σύμφωνα και με παλιότερε τοποθετήσει του, σε προηγούμενες θητείες ε, εργάζεται πολύ εντατικά ε, για την επεξεργασία μιας ε, πρότασης. Το έχουμε συζητήσει με το πολιτικό γραφείο του Αντιπρόεδρου κ. Τίμερμαντς και από ό,τι καταλαβαίνω ο ίδιος και η γενικότερα Κομισιόν δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάρει μια τέτοια πρόταση από εμά και μετά να δει πώς θα τη χειριστεί. Η ερώτηση δική μας είναι εξής. Ε, θα μπορούσατε να πάρετε μέτρα για να στηρίξετε τη θέση του Κοινοβουλίου, την έκκληση του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και την μελλοντική πρόταση του Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Θα θέλατε να μας συμβουλέψετε πώς να προωθήσουμε ένα τέτοιο νόμο. Ασφαλώς κατανοώ ότι υπάρχουν ευαισθησίες μέσα στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Αλλά πιστεύω, μάλλον ανακάλυψα και εγώ σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι ε, υπάρχει μια ένα ευρύ αίτημα, ένα αίτημα που έχει ευρύ υποστήριξη και καλεί τις, ε, τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να καταλήξουν σε ένα κοινό διοικητικό δίκαιο. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς μπορούμε να το προωθήσουμε. Δεύτερον, ο συνάδελφός μου το μίλησε για τις μονοπρόσωπες εταιρείες και όσο πιο πολύ κανείς βλέπει την πρόταση, τόσο πιο πολύ ανησυχεί ότι ε, με το παρόν πλαίσιο εταιρικού δικαίου είναι δύσκολο να καθυσυχαστούν οι αμφιβολίες ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση φοροδιαπηγής ε, ή ε, μαύρης πλαστής εργασιακής σχέσης. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πού βρίσκεται το εταιρικό δίκαιο αυτή τη στιγμή και το πώς αυτό το καινούριο στάτους, το καινούριο καθεστώς μονοπρόσωπης ΕΠΕ θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό. Νομίζω ότι ε, αναφέρθηκε και η οδηγία 14 περί της ε, έδρας των επιχειρήσεων. Κύριε Κέστα, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε για την εισήγησή σας. Θα ήθελα να πω κάτι για τρία θέματα. Πρώτον, όσον αφορά το πρόγραμμα REFIT. Πράγματι, είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας να καταλήξουμε σε μείωση της γραφειοκρατίας. Οφείλουμε όμως να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόμενους να μην αντιμετωπίζονται ως κάτι που μπορεί κανείς να το ρυθμίσει μόνος του. Παραδείγματος χάνει η οδηγία για την ε, ε, προστασία του εργαζόμενου κατά την εργασία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει ε, κάποια εναρμόνιση και θέλω να μας πείτε κατά πόσον θα προσέξετε, θα μεριμνήσετε έτσι ώστε στο πλαίσιο του ΡΕΦΙΤ οι διατάξεις υγείας για την προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της κατάργησης γραφειοκρατίας να μην εξελιχθούν εις βάρος των εργαζομένων ή θέματα κατώτατου μισθού. Μήπως και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές και υπερβολικές διατάξεις. Κατόπιν τίθεται το θέμα της αυτονομίας των συλλογικών συμβάσεων. Αυτά είναι θέματα όπου τίθεται και το πρόβλημα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, εδώ πρέπει κανείς να προσέξει να μην παρέμβει στο θέμα της αυτονομίας των ε, συλλογικών συμβάσεων. Κάτι άλλο που ε, θέλω να ρωτήσω. Έχει σχέση με την έκθεση Ρέντα. Στην Νομική Επιτροπή κατορθώσαμε να επιτύχουμε ευρεία συνένεση που σφραγίστηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να ρωτήσω πώς το βλέπετε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων κυρίως αναφορά την ελευθερία του πανοράματος και Πώς ακριβώς βλέπετε τη σημασία των δημιουργών στην Ευρώπη πάντα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα. Μήπως στο μέλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αν αλλάξουν τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα του δημιουργούν χωρίς βεβαίω να περιορίζεται και η ελευθερία του διαδικτύου. Και το τρίτο αφορά έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με ενδιαφέρει να μάθω κατά πόσον θα προσπαθήσετε κι εσείς έτσι όταν, θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβληθεί και μία ποσόστοση για γυναίκες έτσι ώστε να μην εξακολουθήσει να υπάρχει η κυριαρχία των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Άκουσα με πολύ προσοχή την Επίτροπο. Την ευχαριστώ για την δουλειά που έχει κάνει και ιδιαίτερα για ορισμένα σημεία του προγραμματός της. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο-τρεις πτυχές που μου φαίνονται σημαντικές. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γυναίκα που θέλει να εργαστεί πρέπει να απαρνηθεί τη μητρότητα. Η γυναίκα από την άλλη που θέλει να γίνει μητέρα πρέπει να απαρνηθεί την δουλειά της. Αυτό είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υιοθετηθεί νομοθεσία που θα δημιουργεί ίδιες, τις ίδιες ελάχιστες συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορούν να είναι και μητέρες και εργαζόμενες μαζί. Η εργασία δίνει αξιοπρέπεια και απελευθερώνει τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει έτσι ώστε να εγγυηθεί αυτή την ελεύθερη επιλογή για τις γυναίκες. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένας ελάχιστος, ένας κατώτατος μισθός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μια βάση κάτω από την οποία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αμείβεται ένας Το επίπεδο αυτού του κατώτατου μισθού θα αντιπροσωπεύει την αξιοπρέπεια, το, την ελάχιστη αξιοπρέπεια που μπορούμε να δεχτούμε εμείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι μισθοί θα ισοπεδωθούν. Αυτό θα πρόκειται για ένα ελάχιστο, ένα κατώδος μισθός. Επίσης, ε, ένα, πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσό για διατροφή ε, σε περίπτωση διαζυγίου όταν υπάρχουν παιδιά. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο ποσό διατροφής για τα παιδιά κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται να καθορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία διατροφή. Επίσης, μια ελάχιστη σύνταξη αναπηρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες θα έχουν το ίδιο ποσό. Και πάλι, θέλουμε απλώς κατώτατα όρια προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Τέλος, θα ήθελα να σας ζητήσω να υιοθετηθεί νομοθεσία που θα διευκολύνει τις μονοπρόσωπες εταιρείες. Οι μονοπρόσωπες εταιρείες είναι αυτή τη στιγμή ένας τρόπος να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να εντάξουμε ανέργους ή αέργους στην αγορά εργασίας και θα ήθελα να σας παροτρύνω να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα θα πρέπει να υιοθετηθεί, να θεσπιστεί νομοθεσία που θα κάνει δυνατή την ε, δημιουργία μονοπρόσωπων εταιρεών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις. Θα σας παρακαλέσω κυρία Γιούροβα να απαντήσετε. Dámy a pánové, teď vás budu obtěžovat sluchátky, protože je... Θα σας παρακαλέσω να βάλετε τα ακουστικά σας, γιατί θα μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω τσεχικά και θα τα πω και πιο γρήγορα με την ευκαιρία αυτή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα τη κυρία Ρέγκνερ για το πτωχευτικό δίκαιο. Έχουμε καθορίσει κάποιες αρχές σε σχέση με τις εθνικές διαδικασίες κήρυξης στόχευσης, όχι δεσμοριακά δηλαδή. Υπάρχουν συστάσεις, ε, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές όπως η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, δηλαδή με το ελάχιστο χρηματοδοτικό πρόβλημα να μην καταστρέφεται να μπορεί να δίνεται κάποια βοήθεια τα λοιπά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία ότι μέσα σε πέντε χρόνια τα οι μισές επιχειρήσεις χρεοκοπούν. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτωχεύσεων ε, ημερησίως, 600, 600 πτωχεύσεις ε, στην Ευρώπη τη μέρα. Δηλαδή πολλές θέσεις εργασίας ε, χάνονται και γι' αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε για κάποιες βασικές αρχές. Δεν ζητώ μικροδιαχείριση ούτε αναλυτικούς κανόνες ε, για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας διότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά θα ήθελα να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποιες ε, γενικές αρχές γιατί υπάρχει αυτό το νομοθετικό κενό που πολλές φορές πλήττει τη σταθερότητα των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα περιπτώσει αφαιρεγγιότητας ε, φυσικών προσώπων, υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, στο πρόγραμμα. 5 με 7 χρόνια είναι η όλη διαδικασία ε, αποδέσμευση από το χρέος, ενώ μόνο ένας χρόνος για τις ΗΠΑ είναι το σχετικό διάστημα. Πρέπει να δούμε πώς λύνουν οι Αμερικανοί και άλλες χώρες της Ευρώπης το πρόβλημα για να μειώσουμε τις προθεσμίες αυτές και επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε και τις συστάσεις που δεν εφαρμόζονται ακόμη από όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί πρέπει να τηρούνται οι βασικές αρχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δεν είναι πολλά τα κρατη ακόμη που στηρίζουν αυτήν την οδηγία. Women on Board. Ένα μεγάλο κράτος και τρία-τέσσερα μικρότερα είναι αυτά. Ε, προς το παρόν είμαστε πίσω, αλλά έχουμε καλές επαφές θέλουμε να συζητήσουμε και με τη Γερμανία και με άλλες χώρες για να υιοθετηθούν ε, παράομοι κανόνες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα ταλέντα των γυναικών και να έχουμε μεγαλύτερη πολυμορφία στα ΔΣ, διότι αυτή η πολυμορφία αποδείχθηκε ότι είναι πάρα πολύ αποδοτική και για τη σταθερότητα των επιχειρήσεων στην αγορά. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας βοηθήσετε και εσείς ε, επιμένοντας ε, και στις κυβερνήσεις σας ε, για το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν να δούμε και την τελευταία ε, εκδοχή του κειμένου αυτής της οδηγίας που κάνει λόγο για πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια και για ισορροπία μεταξύ των δύο φίλων. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για ποσό στο 40% παρουσία γυναικών. Τώρα σε ό,τι τα δικαιώματα των μετόχων. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω γιατί ένιωσα μεγάλη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα με την ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, με μεγαλύτερη διαφάνεια, όπου οι μέτοχοι ε, είναι πιο ε, διαφανείς οι διαμοιβές τους, οι αποδοχές τους. Ε. Και έτσι περιορίζονται κάποιες βραχυπρόθεσμες, ε, πολύ ρηψοκίνδυνες συναλλαγές, μια τακτική και ε, ε, μάλιστα συνήθειες κατά το παρελθόν που δημιούργησε προβλήματα. Επίσης έχουμε το θέμα των εκθέσεων αναχώρα, που είναι σημαντικό. Γιατί είχαμε κάποιες φορολογικές αποκλήσεις και παρεκκλήσεις. Το στόχο μας όμως που θέλουμε να προωθήσουμε, ε, ο στόχος που θέλουμε να προωθήσουμε είναι να μην υπάρχει φορά αποφυγή και θέλουμε να ξεκινήσουμε και μία διαβούλευση ώστε να προχωρήσουμε και με ένα άλλο νομοθέτημα και να μην αφήσουμε το ζήτημα αυτό μόνο σε μια οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Θα γίνει ο νόμος και τριμερής διάλογη και σίγουρα θα σεβαστώ και την άποψη των ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει αυτή η διάταξη εδώ, σε αυτό το νομοθέτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία της μονοπρόσωπε εταιρείε. το έχω πει επανειλημμένω. Για μένα υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Αφενός ε, η επιγραμμική online καταχώρηση μιας εταιρείας και το κατώτατο κεφάλαιο ενός ευρώ. Όπως είπε η κυρία Ρέγνερ πολύ σωστά, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Διαμακρόν τα συζητήσαμε τον Ιούνιο όλα αυτά. Μίλησαμε και για την προστασία για να μην υπάρχει κατάχρηση του απλουστευμένου αυτού συστήματος ε, της ε, καταχώρησης της ε, εγγραφής νέων εταιριών. Το Συμβούλιο τελικά ενέκρινε μία κατεμέ αποδεκτή πρόταση, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης, εξακρίβωσης της ταυτότητας του ιδρυτή ή ενός μετόχου που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο όλων αυτών ε, στη χώρα. Επίσης έχουμε την ηλεκτρονική υπογραφή και κάποια άλλα στοιχεία προστασίας για να μην υπάρχει κατάχρηση αυτού του απλουστευμένου συστήματος ε, online καταχώρησης. Η ρίζα του κακού στην οδηγία, οι αλλαγές αυτές των εδρών, ναι πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να συζητούμε και να αξιολόγουμε. Γνωρίζω ότι ορισμένοι από εσά φοβάστε αυτό ακριβώ, δηλαδή το ότι θα υπάρχουν διπλή έδρα ε, σε δύο διαφορετικά κράτη-μέλη. Θέλαμε να μελετήσουμε ε, τους κινδύνους, πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο. Σε κάποια ε, κράτη-μέλη δεν προβλέπεται. Θα πρέπει να δούμε τι εμπειρία υπάρχει και αν υπάρχουν και καταχρήσεις. Ε, στην περίπτωση διπλών εδρών και αν αυτό πραγματικά είναι επικίνδυνο και έχει να κάνει με αυτά τα οποία αναφέρατε, δικαιώματα των εργαζομένων, με ενδεχόμενο φόρο διαφυγής, φοροαποφυγής, ξεπλήματος χρήματος κτλ. κτλ. Θα ξανααναλύσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και ίσως έχετε ε, επισημάνει κι εσείς ότι τον Ιούνιο το Συμβούλιο δήλωσε ότι το πρόβλημα αυτό της διπλής έδρας δεν πρέπει να δεν θέλει να συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία. Αναγνώριση εγγράφων. Στο τελευταίο Συμβούλιο, οπότε και οθετήθηκε η γενική προσέγγιση Κομισιόν θα καταθέσει και ένα νέο σχέδιο με έναν πιο μακροσκελή κατάλογο εγγράφων που θα μπορούν να αναγνωρίζονται. Δηλαδή να προσθεθούν εκεί και έγγραφα που αφορούν τι ιδιωτικέ επιχειρήσει, ιδιωτικέ εταιρείε. Συζητήσαμε και τι ε, μεταφράσει σε πολλέ γλώσσε, ε, τι ε, επίσημε μεταφράσει από αρχαίου μεταφράσει κτλ. κτλ. Βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσω ότι θεωρώ ότι είναι μια αρχή αυτή η οδηγία. Θα ακολουθήσουν πολλέ ακόμη προσπάθειε για μια περαιτέρω απλούστευση και αμοιβαία αναγνώριση των εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται δηλαδή για την αφετηρία ουσιαστικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το φόρουμ για τα δικαιώματα των παιδιών και τι υιοθεσίε. Δεν ανήκουν ε, στι Βρυξέλλε 2. Είναι αρμοδιότητα εθνική Έχουμε τη σύμβαση της Χάγης. Το 93. Και οι συμβαλόμενοι σε αυτή τη ε, σύμβαση πρέπει να σέβονται ό,τι προβλέπεται. Εμείς θα εστιάσουμε στην προστασία των δικαιωμάτων ε, των ε, παιδιών αλλά μάλλον δεν θα ενταχθεί, ενταχθεί το θέμα των διεθνών υιοθεσιών. Σε ό,τι αφορά το ενέο δικτικό δίκαιο. Ο κύριος Τίμερμανς αντέδρασε θετικά. Δεν είμαι κατά, ούτε εγώ. Απλά θέλω να βεβαιωθώ για δύο, τρία, τέσσερα στοιχεία. Δηλαδή, ότι έχουμε την νομική αρμοδιότητα, ότι είναι αυτό εφικτό, δηλαδή να υπάρξει μια διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, ότι είναι και χρήσιμο και εφικτό από πλευρά περιεχομένου. Η δίκηση, η δημόσια δίκηση στα κράτη-μέλη πολλές φορές ε, ε, βασίζεται σε τελείως διαφορετικές παραδόσεις. Υπάρχουν μεικτά μοντέλα. Δίκηση ε, διαχείριση από το κράτο αλλά και από του δήμου κτλ. Είναι πολλές οι διαφορέ. Όπως και στην περίπτωση τη έτσι και εδώ θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν κατάλογο κανόνων που μια δημόσια διοίκηση ε, που θέλει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και υπευθυνότητα θα πρέπει να τηρεί σεβόμε τα δικαιώματα των πολιτών. Άρα δεν είμαι καθόλου αντίθετη, το, το αντίθετο θα έλεγα. Ε, και θεωρώ καλή αυτή την ιδέα και αυτό γιατί στη χώρα μου Έχω περάσει από τα διάφορα στάδια της δημόσιας δίκησης και γνωρίζω πόσο παροχημένοι είναι πολλές φορές οι κανονισμοί, δεν είναι προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες συνθήκες και σίγουρα είναι καλό να γίνει μια ανάλυση και από νομικής πλευράς και σε σχέση με το τι πρακτικές συνέπειες ε, θα ε, υπήρχαν. Καλό να γίνει λοιπόν αυτή η ανάλυση, δεν είμαι αντίθετη, δεν είμαι κατά και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία κάνετε λόγο, σίγουρα θα εμπνεύσει και εμένα προσωπικά. Υπήρχε και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο αφορούσε τις μονοπρόσωπες εταιρείε. Έχουμε μια αναλυτική, μια λεπτομεριακή ανάλυση του εταιρικού δικαίου, του δικαίου επιχειρήσεων και εστιάζουμε στους ε, κανόνες για την ε, Επίλυσε τον συγκρούσεων και για την αρχή του εφαρμοστέου δικαίου. Πρέπει να επιταχύνω από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη. Ο κύριος Κέστν έκανε ένα ερώτημα για την αναδιατύπωση και την προστασία των εργαζομένων. Την οδηγία για το καθεστώς των εργαζομένων, διότι στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης και της αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, των μισθωτών δεν πρέπει να περιοριστούν. Έχω μια γενική παρατήρηση. Εάν σε αυτή τη αναδιατύπωση εξετάζουμε την νομοθεσία, τι βλέπουμε ή τι θα δούμε κυρίως. Θα δούμε αν υπάρχουν ξεπερασμένα, παροχημένα στοιχεία το ευρωπαϊκό δίκαιο με τα οποία δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων και αυτά θα πρέπει να τα διορθώσουμε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Η κυρία Τάισα τουλάχιστον, η αρμόδια επίτροπος, νομίζω έτσι θα προχωρήσει. Για το δικό μου τομέα δραστηριοτήτων, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την πολιτική καταναλωτών, κατά το παρελθόν είχαμε πολλές οδηγίες που ε, σωρεύτηκαν για να ρυθμίσουν ε, συγκεκριμένα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε μήπως ήδη ε, έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα ορισμένες διατάξεις των οδηγιών αυτών και αν χρειάζεται να είναι τόσο πολυάριθμες οι οδηγίες αυτές ή καλό θα ήταν να είναι πιο απλή η νομοθεσία με λιγότερα κείμενα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Θα δούμε επίσης, θα επανεξετάσουμε τις απαιτήσει, τι ανάγκε και θα δούμε και το θέμα τη νομική οικονομία. Δηλαδή θέλουμε καλύτερη νομοθεσία, αυτή είναι η λογική που μας διέπει και αυτό νομίζω ε, είναι και αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έχουμε συνεργασία με τους βουλευτές στο πλαίσιο ιδίως αυτής της άσκησης, της αναδιατύπωσης δηλαδή των σχετικών νομοθετημάτων γιατί θέλουμε να έχουμε feedback, θέλουμε να έχουμε και τη δική σας συμβολή για να αποφασίσουμε ποια νομοθετήματα χρήζουν προσαρμογών, ποια νομοθετήματα πρέπει να καταργηθούν ενδεχομένως ε, και ποια νομοθετήματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες από που φορούν τον κύριο Έτιγκερ και δεν θα παρέμβω. Υπάρχουν τα θέματα των δικαιωμάτων δημιουργού που δεν είναι δικαιωμοδιότητα, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του πανοράματος, δηλαδή το δικαίωμα φωτογράφησης, βιντεοσκόπηση, δημοσίωχο κτλ. Και τα δικαιώματα δημιουργών και των καλλιτεχνών, σίγουρα πρέπει να τα προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά. Αυτή είναι η άποψή μου, η γενική μου άποψη και δεν θα επεκταθώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαστήριο, Φαντάζομαι ότι τα στοιχεία για αύξηση των υποθέσεων ενώπιν του δικαστηρίου είναι ορθά. Σίγουρα θα ε, χρειάζεται αύξηση των δικαστών, ε, φαντάζομαι, και εμπιστεύομαι τα στοιχεία αυτά. Δεν είναι όμως δική μου αρμοδιότητα το θέμα. σε ό,τι αφορά το φύλλο, οι υποψήφοι προτείνονται από τα κράτη-μέλη, υποψήφοι δικαστές. Και οι ορισμοί νομίζω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Υπάρχει συνεχής προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ε, κάναμε μία έρευνα για να δούμε αν υπάρχει ισότητα φύλων ε, στον τομέα της δικαιοσύνης. Και βλέπουμε ότι στα πρωτοδικεία οι περισσότερες είναι δικαστίνες. Ε, όσο ανεβαίνει όμως ε, ο βαθμός κοιοδοσίας, τόσο λιγοστεύουν οι γυναίκες και ε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, ισότητα φύλων. είμαστε στη φάση εκπόνησης ενός νέου νομοθετήματος και μη νομοθετικών μέτρων για να αντικαταστήσουμε στο μέλλον την οδηγία που καταργήθηκε σε ό,τι αφορά την ε, άδεια μητρότητας, ε, τη γονική άδεια. Ε, θέλουμε να αλλάξει η προσέγγιση της γυναίκας ε, ως μητέρας για να έχει όλες τις δυνατότητες επιλογής. Και δεν μιλάω μόνο για τη μητέρα ή για το γονέα. Οι γονείς να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν αν θέλουν να ασχολούνται με τα παιδιά τους ή με τη σταδιοδρομία τους. Και καμία από τις δύο αυτές επιλογές δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον πατέρα ή τη μητέρα να έχει μια ικανοποιητική επαγγελματική και οικογενειακή ζωή και να μπορεί να έχει και μια ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Με την κυρία Τάισεν, την αρμόδια ε, για την απασχόληση επίτροπο συνεργαζόμαστε και μέχρι τα τέλη του έτους θα γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, οπότε και θα καταθέσουμε αυτό το σχέδιο προς διαβούλευση. Υπάρχουν επίσης και μη νομοθετικές δυνατότητες όπως είπα, που αξιοποιούμε. Για παράδειγμα, φέτος έχουμε ε, διατυπώσει πολλές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Θα αναφέρω μόνο ε, το πρόβλημα της ανισομερούς εκπροσώπησης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπήρχαν συστάσεις ώστε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν και στην προσχολική εκπαίδευση, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες δεν μπορούν να εργαστούν ε, γι' αυτό το λόγο. πρέπει να κρατάνε τα παιδιά τους. Και ένα άλλο θέμα είναι η διαφορά στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών, που είναι και αυτό ένα αρνητικό στοιχείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μονοπρόσωπες εταιρείε, και το έτοιμά σας ε, να ασχοληθούμε κατά προτεραιότητα με το θέμα αυτό. Απαντώ θετικά και καταφατικά έχουμε υπόψη μας όλους τους κινδύνους. Έχουμε ε, καταλάβει τη διακυβεύτητα με αυτό το σχέδιο ε, κειμένου, αλλά να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν κάποιος στην Ευρώπη θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση. Αυτό πρέπει να τον θεωρήσουμε αυτήν έναν άνθρωπο που θέλει να απασχοληθεί ο ίδιος αλλά να απασχολήσει και άλλους εργαζομένους και ουσιαστικά να κάνει ένα έργο κοινοφελές ένα έργο ε, κοινοφελές προς την κοινωνία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, βάλουμε εμπόδια στο δρόμο του αλλά να τον διευκολύνουμε. Και Νομίζω ότι πολύ αποτελεσματικά και εύκολα μπορούμε ακριβώς να βοηθήσουμε με την απλουστευμένη αυτή εγγραφή καταχώρηση και με το ελάχιστο ε, μετοχικό κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μαγκίνε, Αντιπρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Καταρχάς ε, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που μου επέτρεψε να συμμετάσχω και εγώ στη σημερινή ακρόαση. Είμαι αρμόδια βέβαια για θέματα διαμεσολάβηση σε περίπτωση απαγωγής ε, παιδιών. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας πω, με μεγάλη χαρά άκουσα που είπατε ότι μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα αυτά προ όφελο του παιδιού και τίποτα άλλο να μην πείτε αυτό μου αρκεί. Βέβαια, ακόμα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά για να πετύχουμε αυτά που είναι προς ε, όφελο του παιδιού. Όπως ξέρετε υπάρχει ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 και προσβλέπουμε στο να συνεργαστούμε μαζί σας για την αναθεώρηση του κανονισμού αυτού. Υπάρχουν πολλά θέματα όπως ε, η ερμηνεία της, ε, ε, του σπιτιού του παιδιού ή η διαφορετική ερμηνεία σε δύο διαφορετικά δικαστήρια, σε διαφορετικά Άλλο, ποιος θα ελέγχει την απόφαση του δικαστηρίου και την εφαρμογή ε, της απόφασης αυτής. Και πίσω από όλες αυτές τις δυσκολίες έχουμε πολύ σεθνά παιδιά τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τον ένα γονιό, έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι τους που το γνωρίζουν και έτσι βρίσκονται κάπου στο κενό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω, εγώ έχω να κάνω με πολλές περιπτώσεις που φτάνουν στο γραφείο μου, μερικές μπορώ να βοηθήσω, σε μερικές σε άλλες όχι. Ε, είναι τεχνοκρατική, γραφειοκρατική δουλειά και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν μια πολύ καλή βάση ε, και μπορούμε και εμείς να σας βοηθήσουμε. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η διαδικασία καθυστερεί, υπάρχει αυτή η έννοια της ε, γρήγορης και αμελητή επιστροφής, αλλά το μόνο που καταφέρουμε σε ορισμένε περιπτώσει είναι να επιστρέψουν τα παιδιά ποτέ όμως γρήγορα και αμελητή όπως είπαμε. Σε κάποια κρατημέλη ο γονιός ε, ταξιδεύει με το παιδί του γιατί ενδέχεται ε, σε ένα κράτος μέλος, αν γίνει εκεί η δίκη, να έχει πιο ευνοϊκή μεταχείριση από ό,τι σε κάποιο άλλο. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να το λάβετε υπόψη στη δουλειά σας. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε ε, μπορώ να ε, τα πω κατηδίαν με την κυρία Επίτροπο σε κάποια άλλη φάση. Θα κλείσω με δύο παρατηρήσεις. Έχει τεθεί το θέμα της ε, υιοθέτηση χωρίς την γονεϊκή συνένεση. Αυτό το εξέτασε η Επιτροπή Αναφορών και το εξέτασε και εγώ και πολλές ε, πρεσβείες ασχολούνται με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε. Εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν διαφορές στα συστήματα κοινωνικής μέρημνας των κρατών μελών. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο καταλήγουμε και σε διαφορετική ερμηνεία του τι είναι προς όφελος του παιδιού. Ε, διαφορετικά ερμηνεύεται η υπόθεση όσον αφορά την ε, χώρα από την οποία προέρχονται οι διάδικοι και την χώρα στην οποία εργάζονται. Πιστεύω πάντως ότι πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου αυτά που είπατε κι εσείς και λέω κι εγώ, αυτό που υπερέχει είναι το συμφέρον του παιδιού. Όχι ή, ε, τα ενδιαφέροντα των γονέων ή ε, το δικαστικό σύστημα. αυτη λοιπόν είναι η τομης όπου κατά την άποψή μου πρέπει να ακολουθήσουν περισσότερες συζητήσεις. Ως ε, διαμεσολαβήτρια ή διαμεσολαβητή, αν θέλετε για υποθέσεις απαγωγής παιδιών. Ε, ήθελα να θίξω αυτά τα θέματα γιατί όσο περισσότερες υποθέσεις έχω στα χέρια μου διαπιστώνω όλο και περισσότερο ότι το σύστημα έχει κενά. Άρα δηλαδή με βάση τις δικές σας προτάσεις εναπόκειται σε εμά τους νομοθέτες να βελτιώσουμε το σύστημα, να λειτουργεί το σύστημα. Πρόσφατα σε κάποια ομιλία σας αναφέρατε ότι υπάρχουν περίπου 60 εκατομμύρια μεικτά ζευγάρια. Άρα δηλαδή το πρόβλημα θα ε, επιταθεί. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, νομίζω επειδή είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να θίξουμε το θέμα αυτό στους ε, εκλογείς μας. Όχι απαραίτητα όταν υπάρχει διένεξη, ε, γενικά σε μια συζήτηση να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες για τα δικαιώματα των παιδιών ε, γιατί ξέρετε είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσει κανείς τα θέματα όταν δεν υπάρχει σύγκρουση γιατί σε περίπτωση σύγκρουσης είναι πολύ δύσκολο για τους άμεσα εμπλεκόμενους να βάλουν τα συμφέροντά τους κατά μέρο και να κάνουν τη σωστή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω. Η κυρία Επίτροπος. Ε, οι Βρυξέλλες 2α ε, έχουν δουλέψει ε, για 10 χρόνια αλλά πρέπει να τροποποιηθούν γιατί και εμείς παίρνουμε ερωτήματα και εσείς αναφορές ε, για γεγονότα στα οποία η σύγκρουση μεταξύ των γονέων βαραίνει τελικά τα παιδιά και τα παιδιά είναι αυτά που πληρώνουν το τίμημα. Για, την πρότασή μας ε, συζητήσαμε με Μακρόν και για παράδειγμα την περασμένη Παρασκευή στο Συμβούλιο. Εκεί όλοι οι υπουργοί ανέφεραν τις δικές προτάσεις ε, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, πώς θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστηρίων, πώς ε, θα εμπλακούν περισσότερο οι αρχές, οι κρατικές αρχές, το, το αναφέρατε και εσείς, και πώς μπορούμε να άρουμε τα εμπόδια έτσι ώστε να επιταχύνουμε την απόδοση της δικαιοσύνης. Πολλές ε, καινούριε και ενδιαφέρουσες ιδέες. Οπότε πήραμε πραγματική ενθάρρυνση και μου δίνετε κι εσείς ενθάρρυνση προκειμένου να επιταχύνουμε. Τώρα θα αναλύσουμε ε, διάφορες πηγές, ε, των εμπειρογνωμόνων, μελέτες, ε, ε δημόσια διαβούλευση και το φθινόπωρο θα περάσουμε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και ελπίζω θα το έχουμε έτοιμο το κείμενο την Άνοιξη από πλευράς κομισιών. Ελπίζω ότι δεν θα εμφανιστούν εμπόδια, διότι όλοι συμφωνούμε. Είναι, νομίζω συμφωνούμε ότι αυτή είναι η σωστή μέθοδο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανεί άλλο να ζητάει το λόγο. Τελειώσαμε και το σημείο 4 λοιπόν. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Αναμένουμε και περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. So, uh, dear colleagues, may invite you... Συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ βάλτε την ε, κάρτα σας στη σχισμή. Um, so you will guide me. can we, Ας ξεκινήσουμε τη we would need a bit more of silence. Παρακαλώ πολύ περισσότερη ησυχία. We begin by the authorization for Ξεκινούμε με την οξιοδότηση της Αυστρίας, Βελγίου και Πολωνίας να ακυρώσουν σύμβαση Λαπέστη για τις συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. I close the vote. Λήξη ψηφοφορίας. Adopted. Uh, we... Υιοθετείτε. Εγκρίθηκε. Περνάμε στο σημείο 9, 30 και 31η ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία σε ΑΦΚΟ 1, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται, εγκρίνεται. Αύκο 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμβη 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμβη 4, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμβη 5, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV8 υπέρ κατά αποχές Πέτει ένα υπέρ κατά αποχές ε, ονομαστική επιβεβαίωση με ηλεκτρονική σοφορία. And it Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αύκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MV1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MV6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. MV7 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση παρακαλώ. this 7 has been adopted. Uh, Εγκρίνεται. 5 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 23 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Adopted. Εγκρίνεται. 526 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Τα αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμβη 10 υπέρ κατά α, ηλεκτρονική βεβαίωση. Adopted. Uh, compromise Εγκρίνεται. Συμβαστική για 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αύκο 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α. Επιβεβαίωση. Ας επιβεβαιώσουμε λοιπόν. Rejected. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σημαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμβη 19 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίνεται αλλά ας κάνουμε μια ηλεκτρονική υπαλήθευση Seems to be. Yes. Adopted. Εγκρίνεται. Σημαντική τροπολογία 8 υπέρ. όχι, συγγνώμη, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Let's check. Not everyone has uh, a Everybody voted. Uh, I closed the vote. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 38-39. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αύκο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αύκο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Λιμπέ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ κατά. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Yes, maybe so, but let's hope there was a majority. No, it. Oh my God. Uh, Απορρίπτεται. Λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε εννέα υπέρ κατά απορρίπτεται. Λίμπε δέκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η Λίμπε 12 υπέρ κατά ε, επανέλεγχος. Ε, η Λίμπε 13 υπέρ κατά εγκρίνεται η λίμπε 13 λίμπε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η λίμπε 16 υπέρ ...ΕΝΒΙ 16 υπέρ κατά έλεγχος απολύτεται Απολιτέτε. 11-17 υπέρ κατά πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος NV17 παρακαλώ Εγκρίνεται. Η 527 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένβι 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ένβι 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε τώρα για την έκθεση στο σύνολό της με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Adopted εγκρίθηκε η έκθεση. Πάμε τώρα στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Amendment 2 in favor. Τροπολογία 2. Ο κύριο Σάια. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ζητήσω το εξή. Επειδή η σημαστική πρόταση 9 δεν καλύπτει την 35, θα ήθελα να υπάρχει μια ξεχωριστή ψηφοφορία επ, αυτού, επ αυτής. Το έχουμε ήδη πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα όμως να επιβεβαιώσω ότι επιθυμώ να υπάρχει ε, ξεχωριστή ψηφοφορία επί της ε, τροπολογίας 35. Η κυρία Κάουφμαν. Μιλήσαμε γι' αυτό, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά συμφωνήσαμε επίσης να ψηφίσουμε πρώτα για τη συμβαστική πρόταση και μετά για την τροπολογία 35. Okay, thank you. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 8 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 13 υπέρ Κατά. ηλεκτρονικό έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 19, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ εγκρίνεται 28 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ εγκρίνεται η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, αφού το θέλετε. Απορρίφθηκε. Η εννέα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πράγματι απορρίφθηκε. Τώρα αυτή την τροπολογία 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Και πάλι ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίθηκε. Πάμε στην 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 40 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίφθηκε. Ας κάνουμε καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 42 υπέρ προφορική τροπολογία ο κύριος Σάια. Είχαμε ελπίσει ότι ε, θα είχαμε μεγαλύτερη αποδοχή και θα προσθέτει τις λέξεις. Μετά την υποβολή στην Επιτροπή όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανισμού. Αυτή είναι η αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε. Πολύ ωραία. Με αυτή λοιπόν την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 43. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 50 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο της ε, γνωμοδότησης εγκρίθηκε με σαφήνεια συγχαρητήρια στην κυρία Κάουφμαν πάμε τώρα στις ενιαίες ψηφοφορίες. Σημείο 11. Ορίστε. Είστε αντίθετοι να ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές τις ε, αναφορές. Όχι. Επομέν, χωριστά. Σημείο 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά The point, single votes point 12. 12. Τα single votes. Κυρία Ρέγκνερ, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι στη λίστα ψηφοφορία είναι λίγο διαφορετική αρρύθμιση. Μας δίνεται ένα λεπτό να το ελέγξουμε και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε. in Ordnung øh, für die Abstimmung am er Block. Danke. Yes, but there has been... Μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ όλε. αλλά κυρία Ρίκνε, λέει ο Πρόεδρος, ε, υπήρξε αντίρρηση προ αυτό από άλλε πολιτικέ ομάδε. άρα πρέπει να ψηφίσουμε μία-μία. Για το 11 να επαναλάβουμε όμω την ψηφοφορία για να μην ε, έχει γίνει λάθο, Ψηφίσουμε το 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία σχετικά με την εντολή για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016. Εδώ έχουμε τρία τμήματα. Είστε όλοι έτοιμοι. Σημείο 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες μας And now we continue. Θα συνεχίσουμε τώρα λοιπόν και κλεισμένων των θυρών Παρακαλώ λοιπόν όλους και όλες όσοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται